αφορά ορισμένου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίε. Ο κύριος Κλίντ, εισηγητή, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρότασή της για ε, αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας ε, σχετικά και δημιούργησε τη βάση των όσων σήμερα συζητούμε. Ήταν το χρονοδιάγραμμα πραγματικά πάρα πολύ φιλόδοξο. Αν θέλαμε να καταφέρουμε κατά τη διάρκεια ακόμα της παρούσης θητείας να έχουμε επιτυχίες ε, και να περάσει αυτή η οδηγία που ήδη από το 1985 υπάρχει στην πρώτη της μορφή. Στόχος για τη μεταρρύθμιση αυτή ήταν να βεβαιωθούμε ότι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου θα αυξανόταν και να ε, έχει τη δυνατότητα να μειώνει το κόστος στο λειτουργικό της να αναπτύξει νέες δυνατότητες και να βεβαιωθεί ότι ε, ο Κάθε ένας που παρέχει τέτοια ε, ταμεία και τέτοιες ε, υπηρεσίες να έχει πρόσβαση παντού χωρίς να μειώνεται η προστασία των επενδυτών. Αντίθετα, θέλαμε να την αυξήσουμε αυτή την προστασία. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα και πρέπει να σας πω πραγματικά ότι είναι αξιοθαύμαστο και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Στη συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα κατορθώσαμε σε αυτό το σύντομο πραγματικά χρονικό διάστημα να φέρουμε σε πέρας ε, το σχέδιο αυτό. Τα επενδυτικά ταμεία δίνουν τη δυνατότητα στους μικροεπενδυτές να επενδύουν μικροποσά με τρόπο διαφοροποιημένο σε χαρτοφυλάκια, τα οποία χαρτοφυλάκια από εκεί και πέρα την χάνουν επαγγελματικής διαχείρισης οι ευρωπαϊκοί αυτοί ε, θεσμοί τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Δεν προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μόνο στην Ευρώπη και πολλούνται, αλλά και σε πολλές ε, περιφέρειες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Ασία, στην Αμερική και έχουν και πολύ μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση. Θα έπρεπε οπωσδήποτε λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία για να προστατευτεί και το υψηλό επίπεδο και το κύρος των επενδυτικών ταμείων. Ήδη και στο παρελθόν δύο φορές αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε η οδηγία, αλλά και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχώρησε με πολύ μεγάλη προσοχή, ξεκίνησε διαδικασία ε, διαβούλευσης με πράσινη βίβλο και λευκή στη συνέχεια και με εντατική ανταλλαγή απόψεων όλων των ενδιαφερομένων φορέων της αγοράς. Ε, συνολικά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έξι μέτρα που εξυπηρετούν τους αρχικούς στόχους που σας ανέφερα προηγουμένως. Εδώ ε, υπάρχει πρόταση ε, για καλύτερη, ε, πιο εύκολη διαχείριση, ένα είδος διαβατηρίου για διασυνοριακές συνεργασίες για να μειωθεί η ανισότητα που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες μέτρα ε, επένδυση δυνατότητα στα λεγόμενα master funds ε, για να μπορεί ένα ταμείο να εντάσσεται εκεί και να τη χάνει τη διαχείριση του μεγαλύτερου. Ε, τέταρτο μέτρο να υπάρχει ένα φυλάδιο ενημερωτικό δισέλιδο μόνο που να αναφέρει τα σημαντικότερα στοιχεία και τις πληροφορίες και investor information λέγεται αυτό για τους επενδυτές και πέμπτο, ε, καλύτερη και πιο εύκολη διαδικασία δήλωσης και κοινοποίησης δηλαδή όταν ένα ταμείο ε, παρουσιάζεται σε μια νέα χώρα και ζητάει ε, άδεια, να μην χρειάζεται καινούργια διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης από την αρχή. Και ε, στα πλαίσια λοιπόν της ε, δημοσιονομικής κρίσης έπληγε και αυτός ο κλάδος της χρηματοπιστωτικής καλύτερα. Ε, χάθηκαν πολλά κονδύλια και εδώ πραγματικά θα πρέπει γρήγορα να αποφασίσουμε για να εξασφαλίσουμε την αύξηση της αξιοπιστίας των ταμείων αυτών και οι μικροί επενδυτές, επαναλαμβάνω, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του σε αυτό το εργαλείο για να μην τη χάσουν, εν Βλέπω ότι ο χρόνος μου ήδη έχει τελειώσει. Γι' αυτό θα ήθελα να περάσω μόνο σε δύο συμπεράσματα τηλεγραφικά. Πρώτον, Συστήσαμε μια ομάδα, όχι εμεί δηλαδή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την ηγεσία του Ντελαροσιέρ, που θα ασχοληθεί με το θέμα τη εποπτείας στην Ευρώπη. Ελπίζω αυτά που θα ε, προτείνουν και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουν επιτέλου να υιοθετηθούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμπεριληφθούν και στην πρόταση. Και δεύτερον, ιδιαίτερα στι συγχωνεύσει τη διασυνοριακέ των ταμείων, διαπιστώνουμε ακόμα ότι ισχύει διαφορετική φορολογική μεταχείριση ανάμεσα σε διασυνοριακέ συγχωνεύσει και εθνικέ αμυγό συγχωνεύσει και εδώ απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθεί να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού για όλους και όχι διαφορετικές μεταχειρίσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μακρύβη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ε, διευκολυνθεί η περαιτέρω διαδικασία με τον τρόπο που έχετε επιλέξει. Οι αγορές τελευταία αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η προσέγγιση που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο Ιούλιο ήταν μια οδός διαβουλεύσεων και άρχισε πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας με τη χρήση της οδηγίας. Με την απλούστευση και την προώθηση διαμεθοριακών χρήσεων με την προώθηση των μηχανισμών αυτών ώστε να μπορέσουν τα ταμεία να υποφεληθούν από οικονομίες κλίμακος. Τα... Οι ενδείξεις είναι θετικές. Έχουμε βάλει και κανόνες για την ανακοίνωση και την διαφάνεια, ώστε όσοι επιθυμούν να επενδύσουν να έχουν στην διάθεσή τους πλήρες και διαφανείς πληροφορίες πριν λάβουν τις σχετικές αποφάσεις τους. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κάνει προσαρμογές στην πρόταση της Επιτροπής για τις συγχωνεύσεις και για την Key Investor Information. Ήταν φιλόδοξη η στόχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να γίνουν σεβαστοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διαδικασίας συναποφάσεως και σχετικά με το διαβατήριο των μέσων αυτών που είναι ένα σημαντικό μέρος, μέρος της ε, προτάσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ε, περίπτωση όπου τα ταμεία δεν είναι παρκώς προετοιμασμένα Είμαι πεπισμένος ότι η απόφασή μας για, τα θέματα αυτά ήταν η σωστή και οι αποφάσεις του Συμβουλίου θα προστατεύσουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Ε, όπως είπα, άρχισε η προσπάθειά μας τον Ιούλιο του 2008. Έχουμε ήδη ένα σύνολο κανόνων που ξεκαθαρίζουν τις ε, ευθύνες για την ροή των πληροφοριών και για την απαραίτητη υποστήριξη στις ε, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Με την αρχική έγκριση, με την περαιτέρω εποπτεία και ενίσχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχεται το συμβαστικό κείμενο. Όμως δεν έχει τελειώσει εδώ η δουλειά μας. Η επιτυχία μας του Management Copy Passport θα εξαρτηθεί και από τη συνέχεια που θα δοθεί. Θα μας δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που θα σημειωθούν. Έχουν επιβληθεί προθεσμίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκφράσει τη την ε, ανησυχία μας για την, ε, δυνατότητα να τηρήσουμε τις προθεσμίες αυτές. θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει το δυνατόν συντομότερο τη σχετική διαδικασία με τη συνεργασία όλων των μερών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας εγκαίρως. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Κλίντς, εισηγητή, και εκφράζω την ικανοποίησή μου για τον ταχύ τρόπο με τον οποίο ε, συνεργάστηκε μαζί μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρώπη μπορεί ε, σύντομα να ανταποκριθεί με την ε, έγκριση, τελική έγκριση της σχετικής νομοθεσίας και τέλος έχω να κάνω δύο δηλώσεις σχετικά με την έγκριση της εκθέσεως. Πρώτον, για, τις, για τη φορολογήση των διαμεθοριακών συγχωνεύσεων. Σε περίπτωση αντιφατικών εθνικών φορολογικών συστημάτων. Θα δούμε τις συνέπειες όταν θα έχει εγκριθεί η πρόταση. Και σε ό,τι αφορά την εποπτεία, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία, η εποπτική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δική μου σύσταση κατέθεση πρόταση για την ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης Τελαροζιέ για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεργασία εποπτείας. Ο κύριος Γκοζές για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψατε μου πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία που έκανε ο εισηγητής και ο οποίος κατόρθασε ε, να επιτύχει μια μεγάλη συμφωνία και που διαπραγματεύθηκε ένα συμβιβασμό ο οποίος είναι ικανοποιητικός. Η Νομική Επιτροπή γνωστοποίησε τις απαρατηρήσεις οι οποίες λήφθηκαν υπόψη. Η αρχική οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ ήταν η βάση για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία. Τον Ιούνιο 2007 τα περιουσιακό στοιχεία αντιπροσώπευαν 6.000 δισεκατομμύρια ευρώ ε, και οι ΟΣΕΚΑ έχουν 75% ε, της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι εσωτερικές εγγυήσεις των ΟΣΕΚΑ εξηγούν την αναγνώρισή τους από τους επενδυτές πέραν του ευρωπαϊκού χώρου αλλά η ρύθμιση έπρεπε να εξελιχθεί για να ευνοήσει την ανάπτυξη αυτών των ταμείων. Οι τροποποιήσεις του 2001 άνοιξαν στους ΣΕΚΑ νέους τομείς επενδύσεων, αλλά άφησαν ορισμένα ε, σημεία ε, δύσκολα, σημεία συμφόρησης. Έχαμε ε, μια πράσινη βίβλο, μια λευκή βίβλο και έχουμε σημαντικές προόδους ως προς την αποτελεσματικότητα με την πρόταση που υποβλήθηκε για την δική μας ψήφο. Η σημαντικότερη πρόοδος είναι η αναγνώριση ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τις εταιρείε διαχείρισης. Οι διατάξεις που προτείνονται θα επιτρέψουν την χρησιμοποίηση των διαβατηρίων αυτών για τις εταιρείε διαχείρισης ενώ θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία για τους επενδυτές. Πρόκειται για ένα πλήρες διαβατήριο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα μέτρα υποπτίας και παρακολούθησης που προτείνονται θα είναι αρκετά αποτελεσματικά ε, για να εξουδετερώσουν, για να διαλύσουν τους φόβους και τις αμφιβολίες. Επίσης υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο τεχνικό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη για τις κοινοποιήσει, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ή ε, για την ομαδοποίηση ε, ταμείων, ε, κονδυλίων και κεφαλαίων με τους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ. Θα έχουμε επίσης καλούς όρους ανταγωνισμού ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την επιφύλαξη ε, των δράσεων που θα πρέπει να υπάρχουν σε φορολογικό επίπεδο όπως είπε και ο εισηγητής για να αποφευθούν οι στρεβλώσεις. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λούλινγκ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Περισσότερο από ποτέ η πρόταση οδηγίας που το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει μου προκαλεί ένα αίσθημα ανάμεικτο βεβαίως ο κύριος Κλίνς ο εισηγητής εδώ και χρόνια έχει κάνει ένα μακρόπνο έργο και διαπραγματεύτηκε με ταλέντο κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και η οδηγία έχει ορισμένες σημαντικές πρόοδους Είμαι για μια καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της συλλογικής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και χαιρετίστηκε από τον κλάδο αυτόν τον ευρωπαϊκό. Αλλά οι συζητήσει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο δεν ήταν ποτέ πλήρω ελεύθερες εφόσον γνωρίζαμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα έπρεπε ορισμένοι συμμετέχοντες να επέμεναν για το διαβατήριο το ευρωπαϊκό ως προ την αρχή δεν έχουμε τίποτα να πούμε, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε η εισαγωγή του διαβατηρίου για τι εταιρείε διαχείριση να συνοδεύεται με τις απαραίτητες εγγυήσει για την παρακολούθηση, την εποπτεία των ταμείων αυτών, διότι υπάρχει λειτουργία εκτός συνόρων. Με λύπη βλέπω όμως ότι το σύστημα είναι όχι μόνο περίπλοκο, αλλά μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους και θα μπορούσε να προσκρούσει γρήγορα σε πρακτικές δυσκολίες που θα βλάψουν τον κλάδο αυτόν κυρίως ε, για τα κεφάλαια που εξάγονται σε τρίτες χώρες Βεβαίως δεν είναι τρομερές αυτές οι δυσκολίες. Σε άλλες εποχές θα έλεγα μόνο ότι μόνο η πρακτική θα μας επέτρεπε να εξαγάγουμε οριστικά συμπεράσματα και να προσδιορίζουμε ποιος έχει δίκιο μεταξύ αυτών που εμπιστεύονται την ικανότητα προσαρμογής των πρωταγωνιστών της αγοράς και αυτών οι οποίοι είναι πολύ πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Δεν αποκλείεται να υπάρξει επιτυχία στο τέλος, αλλά τίποτα δεν εγγυάται αυτήν την επιτυχία. Η επικαιρότητα, το σκάνδαλο Μέιντοφ και οι συνέπειες πάνω ε, στην συλλογική ε, διαχείριση κεφαλαίων ε, δεν μας καθησυχάζει. Αντίθετα, είμαστε ανήσυχη. Αυτός ο κλάδος ε, βεβαίως πλήττεται από την κρίση την χρηματοπιστωτική. Βεβαίως θα χρειαστούν ίσως προσαρμογές μέσα σε αυτό το πλαίσιο βαθιάς κρίσης. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε επιλογές ε, που να διαλύουν την ευθύνη των πρωταγωνιστών όπου να συνεπάγονται μια ε, πραγματική συνεργασία. Ίσως αυτά να μην θεωρηθούν ότι έχουν σημασία. Αυτή η οδηγία είναι ίσως μια οδηγία που θα ήταν ίσως ικανοποιητική σε μια περίοδο όπου δεν θα είχαμε κρίση, διότι είναι κάπως ξένιαστη αυτή η οδηγία. Διότι όλα εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική της. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η βασική λειτουργία των ΟΣΕΚΑ είναι η προστασία των επενδυτών με την διαφοροποίηση των κινδύνων και με αυστηρούς κανόνες. Ψηφίζοντας αυτό το κείμενο ως έχει, χωρίς να ξέρουμε προς τα που οδεύουμε, είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα αυτός ο ταυτισμός δεν προϊονίζεται τίποτε καλό, γι' αυτό θα απόσχω παρόλο που προσυπέγραψα στις τροπολογίες, στις συμβιβαστικές με το Συμβούλιο, αλλά με τις περιστάσεις που έχουμε οι βελτιώσεις δεν μου φαίνονται επαρκείς σε σχέση με τα θέματα αρχής τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε αυτή τη νέα οδηγία ε, για τις ΟΣΕΚΑ. Πρόκειται για μια σημαντικότατη οδηγία και αυτό ισχύει τόσο για το παρελθόν όσο και για το μέλλον. Πράγματι η εξέλιξη υπήρχε σημαντικότατη από την πρώτη οδηγία η οποία ε, ε, θεσπίστηκε πριν από 25 χρόνια. Θα πρέπει να συντονίσουμε τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις και νομοθετικές. Θα πρέπει να ενημερώσουμε όλες αυτές τις διατάξεις για να λάβουμε υπόψη τις νέες απαιτήσει, το νέο περιβάλλον για να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ε, κινητικότητα, μια μεγαλύτερη ρευστότητα και έναν καλύτερο έλεγχο. Η εργασία στην Επιτροπή Επιτροπή διεξήχθη με ικανοποιητικό τρόπο, με καλή συνεργασία, χάρη στον εισηγητή που ευχαριστώ και χάρη στο Συμβούλιο. Ίσως είχαμε συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την χρηματοπιστωτική κρίση και είχαμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη να ανταποκριθούμε ε, με άμεσο και συνεπή τρόπο. Μπορέσαμε να έχουμε μια καλή συνεννόηση και ελπίζω καλά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει για τις εταιρείες διαχείρισης όσον αφορά στον ορισμό του εφαρμοστέου δικαίου είτε πρόκειται για την εταιρεία διαχείρισης ή για το κράτος, ε, πρόκειται για έναν έλεγχο πιο αποτελεσματικό. Η συμφωνία για τα μέτρα που ζητούνται τώρα από την Επιτροπή, αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι τον μήνα Ιούλιο 2010. Και εδώ έχουμε ε, καλή συνεννόηση σε σχέση με τον μηχανισμό της διαδικασίας για τις εταιρείε διαχείρισης, ε, τις επαφές, ούτως ώστε να ξέρουμε πού θα προσφύγει κανείς σε περίπτωση ανάγκη ακόμα και αν η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει την έδρα της στο, σε αυτό το κράτος. Θα μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία ως προς τον έλεγχο με ε, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και της εταιρείας διαχείρισης. Αυτό είναι θετικό και υπάρχουν επίσης και οι συμφωνίες σχετικά ε, και οι συνεννοήσεις ε, σχετικά με τις ε, συγχωνεύσεις και τους απορροφούντες ακόμα και αν υπάρχουν ακόμη διαφορές ως προς τις διαδικασίες είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είχαν προβλεφθεί και σχετικά με την προστασία των καταναλωτών υπάρχει εδώ μια βούληση ε, ισχυρή ότι θα υπάρχει μια αυτόματη ε, διανομή των διαφόρων φυλαδίων των ενημερωτικών επιχάρτου ε, ώστε να υπάρχει καλή ενημέρωση. Σημεριζόμαστε την ανάγκη να συμπληρωθεί ο φάκελος αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ράιν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φιλελεύθερο συνάδελφο κύριο Κλίντς για την εξαίρετη εργασία του. Πραγματικά πιστεύω σε σύντομο χρόνο κατάφερε ο εισηγητή να βρει ένα καλό συμβασμό. Ακόμα και χωρί χρηματοπιστωτική κρίση είναι δύσκολα τα θέματα αυτά στο χειρισμό του και στη διαχείριση γενικότερα. Τα γνωρίζω πολύ καλά διότι έχω εργαστεί σε αυτό το κλάδο στο ΟΣΕΚΑ ε, το 2001. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί αποτελεσματικά η αγορά για τους επενδυτές, τους καταναλωτές. Και τελικά αυτό επιτυγχάνεται νομίζω. Θυμίζω ότι το 2001 η κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη και προφανής. Ήταν ακόμα πριν τη διαδικασία λαμφαλουσή. Πολλά μέτρα ελήφθησαν τότε, αλλά χρειάζεται να ληφθούν και νέα. Είναι σημαντικό να ενισχύεται και η αγορά και η ασφάλεια των επενδυτών, αλλά και η εποπτεία των ε, ΟΣΕΚΑ. Το είπε και ο Επίτροπος ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, γίνεται μεγάλος λόγος για αυτό το ευαίσθητο και λεπτό θέμα του διαβατηρίου για τις εταιρείες διαχείρισης. Ακούσαμε διάφορα ε, σχόλια, αλλά νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση. Είναι καλό να επιμένουμε πάντα στον ανταγωνισμό και στην εξωστρέφεια για να είναι αποτελεσματική μια αγορά και να λειτουργεί σωστά. Και επίσης να είναι καλέ και πληροφορίε που παρέχονται στους επενδυτέ, Να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα τη πληροφορία. Όταν κατακλείζεται κανεί από πληροφορίε, δεν είναι αυτό κατά ανάγκη σωστό και καλό. Αλλά θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι οι επενδυτέ για να ε, παίρνουν τι αποφάσεις του με τα λόγου γνώσεως. Νομίζω ότι βρήκα μια καλή ισορροπία. Η Ευρώπη ε, προφανώ και χρειάζεται εδώ μια καλώ, λειτουργούσα αγορά και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητέ αξίε πραγματικά γνωρίζουν επιτυχία και εκτός της Ευρώπης οι ευρωπαϊκές. Εποφεληθούμε από αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ράιαν για 1,5 λεπτό. Thank you, Mr. President. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κλίντ, τον εισηγητή, για την εξαίρετη πραγματικά έκθεσή του. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να συμφωνήσουν όλοι στο συμβιβασμό και τον συγχαίρω γι' αυτό. Η αναδιατύπωση τη οδηγία αυτή φέρει περισσότερη γραφειοκρατία και μεγάλο βάρος και φόρτο και ορισμένα κράτη-μέλη ανησυχούν. Αλλά από την άλλη νομίζω προστατεύει και τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Όπως ήδη είπαν ε, προλαλήσαντες, μια ανοιχτή αγορά είναι ε, καλή εξέλιξη και θετική και όταν είναι καλά ρυθμισμένη λειτουργεί σωστά. Σήμερα οι χρηματακορές είναι τόσο αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες που χρειάζονται κοινοί κανόνες για ε, τον κλάδο αυτό που είναι πλέον παγκόσμιος στις ε, επενδύσεις. Όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή, αλλά και παγκόσμια ισχύ. Είναι πρωτοφανή φαινόμενα ε, αυτά και θα πρέπει να συνεργαστούμε παγκόσμια για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μεγάλη ευκαιρία διότι εορτάζουμε τη δεκάτη επέτειο της έλευσης του ευρώ που δείχνει από μόνο του πόσο σημαντική είναι η οικονομική συνεργασία και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χώρα μου η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωζώνης. Το κοινό το ενιαίο νόμισμα προσέφερε σταθερότητα σε δύσκολους χαλεπούς καιρούς παγκόσμια ύφεση στη Ιρλανδία. Αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη, δυστυχώς, θα είχαμε σήμερα τη μοίρα της Ισλανδίας. Θέλω να πω στα μέλη του Συμφέν κυρίω εδώ ότι αν είχε περάσει το δικό του τώρα δεν θα ήμασταν στο ευρώ που μα έλεγαν και τότε ότι ήταν οπισθοδρόμηση. Δεν θα ήμασταν στην ΟΝΕ και η οικονομική μα θέση πραγματικά θα ήταν σήμερα σε επίπεδο Ισλανδία. Θέλω να πω σε εκείνου στην Ελλάδα που στρέφονται κατά τη Ευρώπη και απορρίπτουν τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ε, διαχέουν έτσι μεγάλη σύγχυση στα πνεύματα για τι ε, δεχόμενες επιπτώσεις θα πρέπει να σκεφτούν τι σημαίνει οικονομικά αυτό για την Ιρλανδία. Θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη. Αυτό ε, το χρειάζεται και η Ευρώπη και η επιχειρήσει και η οικονομία μας. Σε ευχαριστώ. Um, Ο κύριος Πέρβης για δύο λεπτά. Uh, ευχαριστώ. Παρόλες τις αμφιγνωμίες σχετικά με τον κανονισμό για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε κλπ. Τούτο εδώ το παράδειγμα είναι ένα καλό παράδειγμα κοινή λογική και μετρημένη ρύθμιση του κλάδου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Σκλίντ δούλεψαν όπω έπρεπε και ευχαρίστω θα υποστηρίξω την πρόταση. Τα ο ΣΕΚΑ είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα για τη σκοτσέζικη οικονομία. Είναι σημαντικό μέσο επένδυση για του επενδυτέ όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, υπάρχει το πρότυπο το οποίο εμπνέει και εμά. Ο κύριο Κλίντ περιέλαβε πολλά από τα σημεία που θεωρούσα εγώ σημαντικά όπως η διαφοροποίηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα για παράδειγμα με επαρκή ε, επίπεδα ασφαλείας και κοινή λογικής και κυρίως πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος στην Ευρώπη. Πολλά από τα οσεκά μας είναι πολύ μικρά και κατακαιρματισμένα. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε συγχωνεύσεις των οσεκά αυτών. Εγώ θα ήθελα μάλιστα αυτό να προχωρήσει ακόμη περισσότερο έτσι ώστε οσεκά με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους να μπορούν να συγχωνεύονται ευκολότερα και να προσφέρουν στον επενδυτή πλήρη προστασία και ενημέρωση για τις αλλαγές αυτές. Και τέλος το διαβατήριο διαχείρισης, το οποίο είναι πολύ σημαντική νέα διάταξη που θα επιτρέψει ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και αποτελεσματικότητα, μείωση της γραφειοκρατίας και αυτό βεβαίως είναι προς το συμφέρον του επενδυτού. Άρα η αναθεώρηση θα ωφελήσει τον κλάδο και πιο σημαντικό ακόμη θα αποτελέσει όφελος για τον αποταμιευτή και τον επενδυτή και μάλιστα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Άρα ευχαρίστω υποστηρίζω την, πρόταση του κυρίου, την έκθεση του κυρίου Κλίντς. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κύριε Μπερές, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα για την εργασία σας, τη δέσμευσή σας και την διαπραγματευτική σας ικανότητα. Η ΟΣΕΚΑ είναι τρόπο να το σήμα κατά των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Είναι καλό εξαγωγικό προϊόν. Αλλά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ανισορροπίες, διότι στο κλάδο αυτό έχουμε χώρες παραγωγούς, χώρες καταναλώτριες και διαφορετικές στρατηγικές λοιπόν. Ένας από τους στόχους της αναδιατύπωσης οδηγίας είναι να οργανώσουμε υπό τις συνθήκες αυτές μια πραγματική σωστή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς των ΟΣΕΚΑ. Έχω λοιπόν τα εξής ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, Κάτι που επανειλημμένα ακούστηκε αυτό το ζήτημα του διαβατηρίου διαχείρισης. Και άκουσα τον Επίτροπο να μας ε, λέει ότι φοβάται μήπως δεν προετοιμαστεί καλά αυτό το διαβατήριο. Μα αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θα πρέπει κανείς να έχει τη βούληση να το προετοιμάσει. Και έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν τελείως αποφασισμένος προς την κατεύθυνση αυτή ο Επίτροπος και χαίρομαι για τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έτσι ώστε στην αδιατύπωση της οδηγίας αυτής να ε, υιοθετήσουμε δημιουργήσουμε ένα πραγματικό διαβατήριο διαχείριση που να επιτρέπει στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί υπό φυσιολογικέ συνθήκε. Δεύτερη παρατήρηση. Ε, τι γίνεται με την παρακράτηση. Για παράδειγμα, ε, στην αναθεώρηση της οδηγίας ε, αν υποχρεώνουμε τις ε, τράπεζες να παρακρατούν το 5% των τίτλοποιήσεων που κυκλοφορεί στην αγορά θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα και με ίσους όρους γιατί θα πρέπει οι ίδιοι κίνδυνοι να διαπώνται από τους ίδιους κανόνες. Να υπάρχουν υποχρεώσεις παρακράτησης και εκεί. Τρίτον, τι γίνεται με την εποπτεία. Κανείς εδώ δεν αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητά μας ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εποπτείας. Όλοι περιμένουμε κατ' πρωτοβουλία ε, του κυρίου ε, Μπαρόσο τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας Ζακ Ντελαρουσία. Αλλά έχει έτσι η κατάσταση που δεν μπορούμε να περιμένουμε επάπειρο ε, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των συμπερασμάτων. Και θα πρέπει αυτό να έχει αντίκτυπο και στην εποπτεία μεταξύ των διαφόρων φορέων παραγωγών καταναλωτών ως Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα της εποπτείας εκεί. Και τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με τα φορολογικά ζητήματα και διακυβεύματα, τα είπε και ο εισηγητής και ο Επίτροπος δεσμεύτηκε. Τι κρύβεται πίσω από τα φορολογικά. Ε, ε, προστατευτισμός και θα πρέπει και να το καταγγέλουμε αυτό αλλά και να το ξεπεράσουμε. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει ε, πρωτοβουλίες έτσι ώστε και στους ΟΣΕΚΑ η φορολόγηση να επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών χωρί θεσμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Σταρκεβιτσούτε για ένα λεπτό. Θα ήθελα να πω και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, ο οποίος μπόρεσε να βρει τον καλό συμβιβασμό. Δεν είμαι όμως πλήρως ικανοποιημένος με αυτήν την έκθεση. Πρώτον, επειδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ετοιμάσουν όλη την νομοθεσία ε, στην γλώσσα η οποία είναι η συνήθις. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στα αγγλικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εργασία, την γραφειοκρατική των επενδυτικών ε, εταιριών. Αλλά δεν πρέπει να δώσουμε προτίμηση σε μία γλώσσα, να χρησιμοποιείται μόνο μία γλώσσα. Επιπλέον πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε επιπλέον νομική αβεβαιότητα, πάντως χάρη σε ποια γλώσσα θα δίνουμε ε, πληροφορίες στον καταναλωτή. Πώς θα τον ενημερώνουμε. Πιστεύω ότι η ευθύνη, η εταιρική και οι όροι του ανταγωνισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το να έχει κανείς ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτός θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι δυνατόν να μειωθεί το κόστος για τους επενδυτές και συμφωνώ με τον εισηγητή για τα όσα λέει σχετικά με τις υφιστάμενες προοπτικές. Ε, που θα πρέπει να αντικατασταθούν με ένα έγγραφο το οποίο θα παρέχει σαφείς πληροφορίες στον δυνητικό, στον ενδεχόμενο επενδυτή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στην φορολογία. Πιστεύω ότι η πρακτική ε, εφαρμογή ε, του διαβατηρίου διαχείρισης μπορεί να καταστήσει ε, δύνατον τα χαρτοφυλάκια αυτά ε, να γίνουν διαθέσιμα σε όλη την κοινότητα και αυτό έτσι θα επιτρέψει να καλύψουμε τα κενά ε, στην αγορά. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Εκτιμώ την εργασία που κάνει το Κοινοβούλιο αυτό παρατηρήθηκε εδώ σε όλες τις παρατηρήσεις. Δεν είναι βεβαίως το τέλος της ιστορίας. Πολλά πρέπει να γίνουν στα κρατη που θα έχουν το έργο της ε, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ε, της οδηγίας και μέχρι το καλοκαίρι του 2011 θα πρέπει επίσης να υπάρξουν ε, και οι εθνικοί ελεγκτές και επόπτες για την καλή εφαρμογή του διαβατηρίου. Θα πρέπει να διευκολυνθεί αυτή η εργασία στον τομέα αυτόν τον επενδυτικό της κοινότητας. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Κλίνς για δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και να συμφωνήσω μαζί του ότι όντω δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Ένας λόγος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο έχουμε επιβάλει σύντομες προθεσμίες είναι για να διασφαλίσουμε ότι πράγματι η εφαρμογή δεν θα καθυστερήσει αλλά ότι θα συνεχίσει με ταχύ ρυθμό γιατί βλέπουμε τις αγορές να αλλάζουν, να, αλλάζουν, να τροποποιούνται με ε, ρυθμό καλπασμού. Η σημερινή συζήτηση έδειξε μια διακομματική υποστήριξη υπέρ της ε, συμβαστικής προτάσεως. Εγώ δέχομαι την άποψη της κυρίας Λούλινγκ που είναι κάπως διαφορετική. Είμαι ωστόσο πεπισμένος ότι το μέλλον θα δείξει ότι οι ανησυχίες της, της κυρίας Λούλινγκ δηλαδή ότι ε, το Λουξεμβούργο ως κέντρο ε, χρηματοπιστωτικών ε, δραστηριοτήτων θα χάσει σημασία δεν θα, δεν θα είναι δικαιολογημένη η ανησυχία αυτή. Η κυρία ε, Μπερές εξάλλου έχει δίκιο που λέει ότι πρόκειται πραγματικά για προσπάθεια δημιουργίας της ενιαίας αγοράς και στον τομέα των ε, ΟΣΕΚΑ. Μιλούμε για ενιαία αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη δεν υπάρχει ακόμη αυτή η ενιαία αγορά. Προχωρούμε σε μια νέα και πολύ φιλόδοξη συνεργασία των οργάνων αυτών. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά πρέπει αυτά τα όργανα να μπορούν να συνεργαστούν και σε άλλους τομείς με τρόπο που να προκαλεί εμπιστοσύνη. Και εάν η οδηγία ασκήσει κάποια πίεση ε, προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο το καλύτερο. Τα ε, μέτρα τα οποία έχει αναφέρει ήδη ο Επίτροπος είναι πολλά και πρέπει να ε, προωθηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι αυτό είναι αλήθεια. Ο ίδιος ο κλάδος ωστόσο πρέπει να κάνει να εκτελέσει τα καθήκοντά του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν έχουμε θίξει το θέμα του fund processing διότι αναμένουμε ότι ο κλάδος θα τηρήσει την υπόσχεσή του να ε, ρυθμίσει τα θέματα αυτά από μόνος του χωρίς εξωτερική νομοθετική πίεση. Ελπίζω σύντομα να ανταποκριθεί ή δε θα είμαστε υποχρεωμένοι στο ορατό μέλλον να αναλάβουμε δράση. Εν τέλει, επιθυμώ να ευχαριστήσω όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ιδίω το Συμβούλιο για την συνεργασία και την υποστήριξη, καθώς και τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, ιδίω την κυρία Μπερές, την κυρία Γκοτάρντι και τον κύριο Γκοζές, αλλά και την Άστιτ Λούλινγκ, η οποία με το μαχητικό πνεύμα που την διακρίνει τοποθετήθηκε και σήμερα ε, προς υποστήριξη των ε, συμφερόντων της χώρας της. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 10.